Good morning. Please be welcome. Good morning, my dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Απευθύνομαι στις εθνικές αντιπροσωπείες, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, να καλωσορίσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση για την Europol. Είναι τιμή μου λοιπόν που προεδρεύω αυτή της δεύτερης κοινοβουλευτική διάσκεψης. Να καλωσορίσω και την Υπουργό Εσωτερικό της Φιλανδίας, ε, της Ευρωπαϊκής Προεδρίας δηλαδή, την κυρία Όχι Σάλο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Όχι Σάλο η οποία θα κάνει μια ανάλυση στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και της στρατηγικής που θα ακολουθήσουμε στην ημερήσια διάταξη μέχρι το 2024. Εκπροσωπεί λοιπόν το Συμβούλιο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων Έχουμε λοιπόν, θα έχουμε μάλλον και ένα δεύτερο γύρο μετά από την παρουσίαση αυτή. From the co-chair of this joint parliamentary conference, Mrs. Talviti, representing the Finnish uh, uh, delegation to this uh, parliamentary conference. Thank you. Thank you. Λοιπόν, η κυρία Ταλβίτη έχει το λόγο. Να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Οχισάλα. Ξέρουμε τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ευχαριστώ ε, για την τιμή που μας κάνετε. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν τον λόγο απευθείας στην κυρία Υπουργό. Έχετε το λόγο κυρία Οχισάλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου και τα μέλη της Europol που είναι εδώ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την δυνατότητα που μου δίδεται να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητικές και φυσικά επηρεάζουν και την Ευρώπη. Οι κοινωνίες μας αλλάζουν προσαρμοζόμεθα σε αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας, της δημογραφίας και του κλίματος. Η εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από πολλές πλευρές. Ανάμεσα στις πιο ε, έντονες απειλές είναι οι κοινωνικές συγκρούσεις, η τρομοκρατία, οι κυβερνοεπιθέσεις, όπως επίσης και τα προβλήματα που παρουσιάζει το κλίμα. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα θέματα για την πολιτική. Είναι θέματα τα οποία δημιουργούν προκλήσεις για το σύνολο της ασφάλειας στην Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι καμία από τις απειλές αυτές δεν πρόκειται να αυτοαναιρεθεί αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα αποφασίσουμε να αντιδράσουμε στις ε, ε απειλές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε το σύνολο της κοινωνίας, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια, τις διακρίσεις ε, Νομίζω ότι αυτό θα προλαμβάνει πολλά θέματα στον τομέα της ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμό σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και το κράτος δικαίου. Θα πρέπει να βοηθήσουμε στην επιβολή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, γένους, ηλικίας και φυσικών δεξιοτήτων θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η έλλειψη διακρίσεων να παραμένει κάτι το σημαντικό και όχι το δευτερεύον. Αυτά όλα θα είναι δυνατόν να τα πετύχουμε αν συνδυάσουμε τις πολλαπλές μας ικανότητες και ταλέντα. Προς την κατεύθυνση αυτή η Φιλανδική Προεδρία λοιπόν ξεκινάει μια συζήτηση για την μελλοντική κατεύθυνση της εσωτερικής ασφάλειας στην Ένωση. Βασικό στοιχείο είναι η βελτίωση της λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου όπως και ο σημαντικός ε, ε, ρόλος υπηρεσιών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων όπως η Europol. Η συνεργασία μας θα βασίζεται σε αποτελεσματικά συστήματα ενημέρωσης, πληροφόρησης και τεχνολογίας και διαλειτουργικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία με πιο λειτουργικό τρόπο. Ε, υπογραμμίζει η Φιλανδική Προεδρία ότι κάθε φάση αυτής της αλήσου της ε, ποινική δικαιοσύνης έχει σημασία μεγάλη και για την δικαστική συνεργασία. Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στον τομέα αυτό θα πρέπει να εξεταστούν με πάρα πολύ προσοχή. Η κλιματολογική κρίση είναι φυσικά η μεγαλύτερη ευθύνη και ευκαιρία των εποχών μας. Η κρίση αυτή ξεπερνά, αν θέλετε, ε, τα θέματα τα παραδοσιακά με τα οποία ασχολείται η πολιτική και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις σε όλα τα μέτωπα και στην ασφάλεια. Πολλά μένει να γίνουν. Υπάρχει μόνο ένας πλανήτης και πρέπει να τον καταστήσουμε βιώσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε το μέλλον να είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει διεθνή συνονόηση. Όπως η Ursula Φοντεν Λάιεν είπε, η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει η πρώτη ουδέτερη κλιματολογικά ήπειρο στον κόσμο το 2050. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε από κοινού τις αποφάσεις που πρέπει. Θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να δράσουμε σε όλα τα μέτωπα έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν στον πλανήτη αυτό. Οι νέοι της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο ζητούν να αναλάβουμε δράση. Εμείς οι ενήλικες έχουμε την ευθύνη να δράσουμε τώρα. Οι νέοι θα πρέπει επίσης να δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία κάνουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και στον τομέα της ασφάλειας γιατί τίποτα δεν οδηγεί στην βίαιη ριζοσπαστικοποίηση από την απώλεια ελπίδα σε ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτείται να καταπολεμήσουμε την κλιματολογική κρίση με φιλόδοξες πολιτικές σήμερα και όχι στο μέλλον. Στρεφόμενοι στο μέλλον τώρα να πω ότι οι ικανότητες που έχουμε για την αντιμετώπιση των λεγόμενων υβριδικών απειλών θα πρέπει να ενισχυθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών. Οι εσωτερικοί παράγοντες στον τομέα της ασφάλειας θα αυξήσουν την αντοχή των κοινωνιών και θα βοηθήσουν την αντίσταση απέναντι σε δυνατότητες επηρεασμού. Η κοινωνική συνοχή είναι το καλύτερο αντίδετο ε, ενάντια σε αυτές τις υβριδικές απειλές που έχουν σαν στόχο την αποσταθεροποίηση των εθνών μας. Πρέπει να δράσουμε από κοινού με διαθρωμένο και συντονισμένο τρόπο. Ο αριθμός των τρομοκρατικών ενεργειών έχει μειωθεί με τα τελευταία χρόνια, αλλά η απειλή της τρομοκρατίας πάντα παραμένει. Η Φιλανδική Προεδρία υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της συζήτησης για την πρόληψη του βίαιου εκτρεμισμού και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το φαινόμενο των ξένων πολεμιστών και η τζιχαντιστική ιδεολογία είναι μια απειλή πάντα για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι η τρομοκρατία υπάρχει και παίρνει πάρα πολλές μορφές και η τρομοκρατιστική απειλή και από πλευρά της βίαιης άκρας δεξιάς δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ταυτόχρονα η πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι δύο αλληλοστηριζόμενες προσπάθειες. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να εδράζονται σε μια συνολική αντίληψη για την ποιότητα και την ταυτότητα των απειλών και την έρευνα γύρω από αυτές. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρόληψη του μίσου συνεισφέρει στην πρόληψη του εγκλήματος και του εξτρεμισμού. Η Φιλανδική Προεδρία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πρόληψη του εξτρεμισμού, ε, του βίαιου εξτρεμισμού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις νέες αναδιόμενες απειλές από τη μία νέες τεχνολογικές μορφές προόδου έχουν βελτιώσει τα ψηφιακά μέσα που έχουν οι αρχές ε, για να προλαμβάνουν και να ερευνούν τις δραστηριότητες της ποινικά κολάσιμες. Από την άλλη η χρήση του διαδικτύου, τα ε, μέσα ε, τα οποία χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς και άλλους παράνομους λόγους αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και το περιεχόμενο το τρομοκρατικό online έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο παρελθόν στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο η Φιλανδική Προεδρία θα συνεισφέρει στην προώθηση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για να τεθεί τέλος στην διάδοση του περιεχομένου του τρομοκρατικού online απαιτείται ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση και πλήρη συνειδητοποίηση των ευθυνών και των καθηκόντων κάθε εταίρου. Εξετάζοντας τα μέσα πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού έχει σημασία να δούμε ότι οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν και όλα τα μέσα μετακίνησης για να προλαμβάνουμε και να ερευνούμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλα τέτοια εγκλήματα, θα πρέπει επίσης ε, να δούμε τι δυνατότητες μας παρέχει το λεγόμενο PNR και σε άλλες μορφές ταξιδίου και μετακίνησης και όχι μόνο στις αερομεταφορές η διεύρυνση της συλλογή των στοιχείων PNR ε, και στην ε, ναυτιλία ε, και επίσης στις διαμεθοριακές οδικές μεταφορές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Όπως είπαμε, τα μέσα μετακίνησης και η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης έχουν επιταχυνθεί στον 21ο αιώνα η παραπληροφόρηση και ο επηρεασμό της ενημέρωσης παίζουν ένα σημαντικό και περίπλοκο ρόλο. Οι τεχνικές παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι ε, καταχρηστικές ε, μορφές ε, παρουσίασης βίντεο, όπως επίσης παραποίηση επίσημων δεδομένων και κλοπή πληροφοριών. Ε, ένα σημαντικό θέμα φυσικά είναι η μορφή της διάδοσης αυτής της παραπληροφόρησης. Ε, συμπληρωματικά απαιτείται δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας. Η Φιλανδική Προεδρία υπογραμμίζει τον ρόλο της Europol και άλλων ευρωπαϊκών υπηρεσιών στην ταυτοποίηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών σχετικών με την παραπληροφόρηση και επηρεασμό ενημέρωσης. Τα φαινόμενα της α, ρητορικής μίσους είναι κάτι το οποίο πέρασε από τις πίσω σελίδες του ίντερνετ στην καθημερινότητά μας. Στα πλαίσια της προσπάθειας επηρεασμού της ενημέρωσης, το φαινόμενο στόχευσης κυβερνητικών επισήμων έχει γίνει κάτι το πολύ κοινό. Ο στόχος της στόχευσης αυτής είναι η παρέμβαση και η διατάραξη των εργασιών των δημόσιων αρχών, η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης του κοινού στους κυβερνώντες και ε, δημιουργία νέων κοινωνικών διπόλων. Η υπογράμμιση ακριβώς ε, της ε, υπονόμευσης της εμπιστοσύνης του κοινού επηρεάζει αρνητικά την ίδια τη δημοκρατία και τις δομές της και τις δομές του κράτους δικαίου. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Μια κοινωνία στην οποία οι αρχές δεν γίνονται σεβαστές, τότε είναι μια κοινωνία στην οποία οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον αντιμετώπιση της ρητορική μίσους είναι κάτι το οποίο έχει σχέση και με την προάσπιση των αξιών των κοινωνιών μας. Παρά την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων, οι πολιτικοί εταίροι θα πρέπει να είναι σε θέση να προωθούν και να διατηρούν την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ανοιχτές και διαφανείς μορφές επικοινωνίας για να μειώσουμε την αποσπασματοποίηση των κοινωνιών μας. Πάντα όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι. Η ελευθερία του λόγου ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Πέραν αυτού η ελευθερία έκφραση συνοδεύεται και από ευθύνες η άλογη αμφισβήτηση των θεσμών των κεντρικών της κοινωνίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και τα πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να ανοικοδομηθούν καταστρέφονται. Προχωρώντας λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που δημιουργούν και οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι νέες αναδυόμενες απειλές. Είναι σημαντικό να εντοπίσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες. Η Φιλανδική Προεδρία υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης της κυβερνοασφάλειας για την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας. Η καταπολέμηση των κυβερνοεκκλημάτων και των κυβερνοαπειλών απαιτεί πόρους, δυνατότητες τεχνολογικές, και ε, ταχύτατη αντίδραση από πλευράς των αρχών. Είναι σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια αυτά ε, τα ηλεκτρονικά στοιχεία να αποθηκεύονται και να δίδονται το ταχύτερο δυνατόν στις αρχές επιβολής του νόμου. Θα πρέπει <coughs> εδώ να γίνει βέβαια αυτό, αλλά να ε, γίνει σεβαστή και η εθνική ε, ακαιρεότητα αν θέλετε των κρατών μελών όπως επίσης και κυρίως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων. Η ε, τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση επηρεάζουν και συνοδεύουν την εσωτερική αγορά και τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να συνοδεύουν τις εξελίξεις αυτές έτσι ώστε η κατοχή των ε, πιο προχωρημένων μέσων να είναι χρήσιμη θα πρέπει οι αρχές επιβολής του νόμου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν και στα πλαίσια ενός δικτυακού περιβάλλοντος 5G, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει το 5G ε, στην εσωτερική μας ασφάλεια. Η Φιλανδική Προεδρία υπογραμμίζει την ανάγκη επανεξέτασης της ισχύουσας νομοθεσίας και της βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και του 5G. Η διασφάλιση λοιπόν της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσής μας, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι βασικό στόχος της Φιλανδικής Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση και πρέπει να είναι μία ένωση αξιών, κοινών αξιών. Είμαστε φιλόδοξοι, είμαστε πολλαπλοί και δεν αποκλείουμε κανέναν σχετικά με τη μετανάστευση και την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουμε, πρέπει να έχουμε μια συνολική στάση που να αντιμετωπίζει και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πλευρές της μετανάστευσης. Είναι κρίσιμο να συνεργαστεί η συνεργασία με χώρες εκτός της Ένωσης και η προώθηση μέτρων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και στο εσωτερικό τους βέβαια. Η Φιλανδική Προεδρία θα κάνει προτάσεις προληπτικών μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης. Η Φιλανδία θέλει να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και την Αφρική. Με τα πολλαπλά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και τον διεθνή μας ρόλο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες πλευρές της μετανάστευσης ε, καλύτερα από ό,τι κάθε χώρα ξεχωριστά. Πρέπει να καταπολεμήσουμε και τους εμπόρους επίσης ε, των μεταναστών και θα πρέπει ε, να δίνουμε το άσυλο εκεί που χρειάζεται και να βελτιώσουμε την κατάσταση των προσφύγων που είναι ήδη στην Ευρώπη. Όπως είπε επίσης η κλιματολογική κρίση είναι βασική απειλή για την εσωτερική μας ασφάλεια. Αυτό είναι προφανές κυρίως ε, στα πλαίσια των συνεπειών της υποχρεωτικής μετανάστευσης και από ό,τι φαίνεται τέτοιες συνέπειες θα έχουμε περισσότερες στο μέλλον. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά λοιπόν την σημασία της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Το πώς θα πετύχουμε θα έχει μείζονες συνέπειες γενικότερα στις υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες αιτίε που προκαλούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση όπως τα δημογραφικά και την ανεργία των νέων. Απαιτείται ένα σωστός τρόπος ανάληψης ευθυνών. Είναι κοινό συμφέρον όλων μας να έχουμε σωστές εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες προέλευσης και χώρες διέλευσης, έτσι ώστε να μειώσουμε τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται και να προωθήσουμε ασφαλείς και τακτούς τρόπους μετανάστευσης. Σχετικά με τη συνολική αντίληψη και τη διασφάλιση της περιοχής Σέγγεν, πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις οδούς της μετανάστευσης και να γνωρίζουμε το πού δραστηριοποιούνται. Ε, μια λειτουργική βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική για το άσυλο είναι σημαντική για το μέλλον της Ένωσης και για την αξιοπιστία και αποδοχή των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε νόμιμους τρόπους μετανάστευσης όπως και ε, επανεγκατάστασης ε, σε σχέση με τα συστήματα των ποσοστώσεων τα οποία λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις όμως. Υπάρχει επίσης ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού συστήματος χορήγησης ασύλου. Αν θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί καλύτερα και σε τακτικές εποχές, αλλά και σε εποχές κρίσης και υψηλής μεταναστευτικής πίεσης. Πρέπει να προχωρήσουμε σε συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις του συστήματος και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η συζήτηση για τη μετανάστευση έχει συγκεντρωθεί κυρίως στα θέματα αλληλεγγύης και σωστού διαμοιρασμού του βάρους, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία για τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος να συνεχιστεί. Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι για τις ε, μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις έχουμε ανάγκη επίσης ε, και για ε, πρακτικά συστήματα υποδοχής μετά από έρευνες και διασώσεις. Η πρόληψη επίσης της απώλειας ζωής, ιδιαίτερα στη θάλασσα, είναι καθοριστικό για μας, δεν βασίζεται μόνο σε νομικές υποχρεώσεις αλλά και σε κοινέ αξίες, προστασία της ανθρώπινης ζωής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε σχέση με την προστασία των απειλών αυτών δεν πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός. Ο σεβασμός των, θεολι... θεμελιωδών δικαιωμάτων και η νομική προστασία θα βελτιώσουν και τις ε, ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του επαναπατρισμού είναι κάτι το οποίο θα ε, περιγραφεί σωστά στην αναθεώρηση της οδηγίας που ισχύει για την ε, επιστροφή των πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα προέλευσής τους. Η χρησιμοποίηση κινήτρων για τέτοιου είδους αναχωρήσεις ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί. Η Φιλανδική Προεδρία επίσης θα πρέπει να φροντίσει, πιστεύουμε, και τις συνθήκες επιστροφής αυτών των ε, μεταναστών. Σχετικά με την προστασία των ε, συνόρων ε, για τη μετανάστευση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να ολοκληρώσουμε επίσης και τον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά σύνορα και την ακτοφυλακή η εφαρμογή του κανονισμού αυτού είναι μια σημαντική κοινή προσπάθεια για την Ευρώπη και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά. Μετά από τη συμφωνία για μια πιο ισχυρή εντολή, η Frontex έχει καλύτερες δυνατότητες για να βοηθάει τα κράτη-μέλη και να βελτιστοποιεί την διαχείριση των συνόρων στην Ευρώπη. Οι επικοινωνίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εύκολες, ταχείες και αποτελεσματικές. Πολλοί κανονισμοί για τα ευρωπαϊκά συστήματα ενημέρωσης έχουν υιοθετηθεί και ενημερωθεί πρόσφατα. κινούμενοι προς το μέλλον θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στη σωστή διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας σχετικά με τις προτάσεις ε, για κανονισμούς που να συμπληρώνουν την ανταλλαγή στοιχείων ε, για τα συστήματα ε, επίσης ATAS, ενημέρωση και αδειοδότηση. Θα πρέπει η Φιλανδική Προεδρία ελπίζουμε να οδηγήσει στην εκκίνηση τριμερών συζητήσεων, τριμερούς διαλόγου μια πλήρως λειτουργούσα περιοχή Σέγγεν, ένας πλήρως, δηλαδή ένας χώρος Σέγγεν ο οποίος να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση είναι κίνητρο ε, για την ευημερία, την ασφάλεια και την ελευθερία στην Ένωση. Η τροπολόγηση του κώδικα Σέγγεν σχετικά με τα εσωτερικά σύνορα είναι κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί σε σχέση και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νέες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελευθερίας δράσης των κρατών μελών. Η Φιλανδία θα αναζητήσει νέες λύσεις για την κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων. Στρεφόμενη στο μέλλον, η Φιλανδική Προεδρία έχει σαν στόχο την εφαρμογή της λεγόμενης ενιαιοποιημένης διαχείρισης των συνόρων. Ε, υπηρεσίες όπως η Frontex παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν τη βασική ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά και διαφανή μέσα, διασφαλίζοντας ότι οι υποχρεώσεις του Σέγγεν γίνονται πλήρως σεβαστές σε σχέση κυρίως με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η Προεδρία της Φιλανδίας θα υποστηρίξει την ανάπτυξη συστημάτων ποιοτικού ελέγχου προωθώντας επίσης ε, την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων είναι βασικός μας στόχος. Η χρηματοδότηση θα καλύψει τις ανάγκες και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ε, της μετανάστευσης, θα προωθήσει νόμιμους οδούς, ε, νόμιμες οδούς μετανάστευσης και θα προλαμβάνει τις παράνομες, τις μη θα έλεγα νόμιμες μορφές ε, ε, μετανάστευσης. Η καταπολέμηση ε, διαμεθοριακών μορφών εγκληματικότητας, τρομοκρατίας και βίαιου σβησοσπαστικοποίησης είναι ένας άλλος στόχος μας. Οι ανάγκες των θυμάτων των εγκλημάτων αυτών θα πρέπει να καλυφθούν. Είναι σημαντικό τα θεμελιώδη δικαιώματα να παραμείνουν σεβαστά και στα πλαίσια αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Κλείνοντας, θα πρέπει να βλέπουμε μακριά όταν πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις για τις πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Ίσονες αλλαγές και, μη, πρόθεσμα προγράμματα δεν αρκούν. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις σοφές οι οποίες να έχουν μέλλον, να είναι μακροπρόθεσμες. Θα πρέπει να το κάνουμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο, με συνοχή, ισχύ και ένωση και εσωτερικά και κανένας δεν θα μπορέσει να μας απειλήσει και να μας διαιρέσει από το εξωτερικό της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό και τώρα να ξεκινήσουμε την αλλαγή απόψεων χρόνος ομιλίας, δύο λεπτά κατά ανά το όριο. Και στο τέλος ε, θα απαντήσει η Προεδρία. Ο κ. Απέλ, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω πολωνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. για την ομιλία αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα για την κυβερνοασφάλεια και τις κυβερνοαπειλές, γιατί προφανώς αποτελούν ένα τεράστιο θέμα στη σημερινή μας ζωή. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία μας. Στην αρχή κάποιος ανακαλύπτει κάτι το οποίο όλη η κοινωνία το χρησιμοποιεί και μετά βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν κινδύνους. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας αυτό που είχε πει ο Orwell δεν θα χρειάζεται να υπάρχει το Υπουργείο Αλήθεια, το οποίο θα λογοκρίνει το διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε το διαδίκτυο. Και θα πρέπει από μόνο του να περιορίζει το διαδίκτυο κακέ πρακτικέ, όπω για παράδειγμα η διάδοση παραπληροφόρηση και επικίνδυνων ιδεών. Αυτό συχνά αποτελεί επιρροή τρίτων χωρών που δεν ενδιαφέρονται ούτε για την ευρωπαϊκή δημοκρατία ούτε για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι στην ε, καταπολέμηση των εξωτερικών αυτών απειλών στο διαδίκτυο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και σταθεροί. Να προσέξουμε λοιπόν να μην δημιουργήσουμε τελικά ένα Υπουργείο Αλήθειας όπως έχει προβλέψει ο κ. Ορουέλ από την Κύπρο. Δεν ακούσαμε καλά το όνομα το οποίο ανέφερε η πρόεδρος. Ε, κυρία Υπουργέ, στην ομιλία σας σήμερα είπατε ότι μία από τις προτεραιότητες της τρέχουσας Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κατοχήρωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και των πολιτών της από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις και απειλές. Αναφέρατε πως αυτός είναι ο λόγος που η Προεδρία ενθαρρύνει και προωθεί δημόσια συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν γνωρίζετε, η πρόταση για επέκταση των αρμοδιοτήτων της νεοσυσταθήσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση της διασυνοραϊκής τρομοκρατίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναφορά σας για την ελευθερία της έκφρασης, πολλές φορές και το ξέρετε, η ρητορική μίσους εντάσσεται από επιτίδιους στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης. Η ελευθερία του λόγου δεν εξυπακούει οπωσδήποτε ασυδοσία και πρέπει όλοι να αντιταχθούμε στεναρά στις ακραίες πολιτικές που βρίσκουν καταφύγιο στο μίσος, στο ρατσισμό και στις διακρίσεις. Σας ευχαριστώ. Thank you. And then Mr. Ευχαριστώ. Κύριε Σοραλέχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την ομιλία σας η οποία ήταν εξαιρετική. Το διαδίκτυο αναμφίβολα έχει γίνει ένα νέο πεδίο εγκληματικής δραστηριότητας και δημιουργεί πολλές προκλήσεις. Υπάρχει μεγάλος βαθμός ασυλίας στις στον κυβερνοχώρο και δεν μιλάμε μόνο για τρομοκρατικές δραστηριότητε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Υπουργέ για το γεγονός ότι αναφερθήκατε στην ανάγκη πρόληψης της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η δραστηριότητα αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες μας και πλήττει άμεσα τους πολίτες μας αλλά και συνολικά τις ε, κοινωνίες μας, ακόμη και το ηθικό των κοινωνιών μας και την ψυχολογία, τη συλλογική, όταν διαδίδονται τέτοια αφηγήματα μίσους. Οπότε η πρόληψη πραγματικά είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα την άποψή σας για δύο θέματα. Θα γνωρίζετε βεβαίως τις ανησυχίες που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό διαφόρων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη γι' αυτό και τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία προκειμένου να, εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Και δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε ποια μέτρα πρόληψης σκοπεύετε να λάβετε σχετικά με το κυβερνοέγκλημα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία σας με τεχνολογικές εταιρείες και τι σκοπεύετε να κάνετε για να επεκτείνετε την συνεργασία σας αυτή. Ευχαριστώ κύριο Μετσού από το Βέλγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Οχισάλο για την ε, σαφέστατη ομιλία σας. Ένα από τα στοιχεία που αναφέρατε είναι το Μητρό των Ονομάτων των Επιβατών, το PNR. Ξέρετε ότι εδώ και πέντε χρόνια περιμένουμε να θεσπιστεί η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Στο Βέλγιο έχουμε έναν ευρύτερο νόμο που δεν καλύπτει μόνο τις ε, αερογραμμές, τις αεροπορικές μεταφορές, αλλά και τις σιδηροδρομικές ε, και άλλες ε, μεταφορές. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων κοινοποίησης τέτοιων δεδομένων, ονομάτων επιβατών, ε, στις εταιρείε. Εσείς τι πιστεύετε, θα πρέπει αυτό να οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θεωρείτε ότι το θέμα αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χεϊνάλαμα από τη Φιλανδία. Thank you, speaker. Uh, and thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Υπουργέ, όχι σ' άλλο, για την εξαιρετικά σαφή παρουσίαση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να, ζητήσω, να ρωτήσω την ε, Υπουργό σχετικά με το ζήτημα της ιδιωτικότητας και των ε, δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι τα δικαιώματα ιδιωτικότητας δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτιδα δύναμη όσον αφορά την προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών της. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο και σαφές ερώτημα στην Υπουργό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και εκτός της Ένωσης, για παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Ευχαριστώ η κυρία Κάνκο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Θέλω να θέσω ένα ερώτημα, βάζοντας όμως και ένα σχόλιο. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ουσιώδεις συζητήσει για ζητήματα που ε, έχουν σημασία. Ξέρετε, από εκεί που κατάγομαι εγώ μπορεί κανείς να χάσει τη ζωή του για τις απόψεις που έχει. Νόμιζα ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαμε δικτατορίες. Όταν όμως ξεκίνησα τη ζωή μου εδώ στην Ευρώπη και μπήκα και στην πολιτική, διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να έχεις μια ουσιώδη συζήτηση, να κάνεις μια ουσιώδη συζήτηση και πολλές φορές τελικά διαπιστώνω ότι και στην Ευρώπη ε, ε χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους διότι έχουν συγκεκριμένες απόψεις. Σαρλί Αντό, για παράδειγμα. Ε, ή υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται, η Σαντιχαλή για παράδειγμα που κρύβεται στη ΣΥΠΑ ακριβώς γιατί είχε συγκεκριμένη άποψη. Υπάρχει και ε, η αρχισυντάκτρια του Σαρλί Εμπντό που δυστυχώς χρειάζεται αστυνομική προστασία λόγω των απόψεών της. Οπότε, Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε για την ελευθερία του λόγου. Θέλω όμως να εστιάσουμε στο γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατον τελικά να κάνουμε συζήτηση στην Ευρώπη για ζητήματα τα οποία έχουν ουσία, που είναι σημαντικά. Και νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η Ευρώπη που εγώ περίμενα να δω. Πώς θα κάνετε εσείς, πώς θα εξασφαλίσετε εσείς οι άνθρωποι να έχουν τα δικαιώματα στην ελευθερία του λόγου τους όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πραγματική ζωή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίρτσικ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ... Εδώ, εδώ είμαι. Με βλέπετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ συνεπτική αξιολόγηση της κατάστασης. Δύο θέματα θέλω να αγγίξω. Το ένα σε ό,τι αφορά την περιοχή Σέγγεν, χαίρομαι που αναφέρετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι οι προκλήσεις μιας ε, περιοχής Σέγγεν η οποία λειτουργεί πλήρως. Και ξέρουμε ότι αυτό δεν αποτελεί μόνο πρόκληση σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν, αλλά και σε ό,τι αφορά τους συνεχιζόμενους εσωτερικούς ελέγχους που γίνονται από διάφορα κράτη-μέλη. Κάνατε δήλωση ότι η Φιλανδική Προεδρία σκοπεύει να προτείνει μια σειρά προτάσεων που μπορεί να ξεπερνούν αυτά που έχουμε μπροστά μας στην παρούσα φάση. Με ενδιέφερε πολύ αυτό και θα ήθελα να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν θέλετε. Πώς μπορούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και πιο γρήγορα να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η εσωτερική έλεγχοι στα σύνορα του Σέγγεν, οι οποίοι είναι παράνομοι, θα σταματήσουν. Δεύτερο θέμα. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με διάφορους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση στο διαδικτύο. Σταθήκατε πολύ στο πώς ε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε το περιεχόμενο, το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδικτύο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που αναφέρω είναι ακόμα πιο βαθύ πρόβλημα, γιατί δεν βλέπουμε τα συμπτώματα καθημερινά ανά πάσα στιγμή είναι κάτι το οποίο το κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του. Άρα ποια είναι η προτινόμενη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την ε, επικοινωνία με τις μεγάλες πλατφόρμες και τους μεγάλους παρόχους του διαδικτύου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση, τη σωστή και έγκαιρη καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελευταίος ομιλητή σε αυτό το γύρο, ο κ. Κάλε, από τη Σλοβενία. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Υπουργό και τους συμπρόεδρους. Συμφωνώ ιδιαίτερως με την παρουσίαση που έδωσε η Φιλανδική Προεδρία υπογραμμίσατε πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα στην παρούσα φάση. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μία λεπτομέρεια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της απληστίας απληστία σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε ό,τι αφορά τα παιδιά μας. Όπως ξέρετε σήμερα, οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει ένα λογαριασμό στα social media και να έχει πρόσβαση μέσω ενός smartphone. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνει κλικ στην επιλογή αν των 18 και οι πολυεθνικές προφανώς δεν τα ελέγχουν όλα αυτά και έτσι βρισκόμαστε με παιδιά 10-11 χρονών τα οποία προφανώς είναι εύπιστα. Και οδηγούμαστε έτσι σε πολλές περιπτώσεις κατάχρησης τέτοιων ε, προφίλ ε, στα μέσα δικτύωσης. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Οριζό, για να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις, ε, οι οποίες θα απευθύνονται στην ε, συνάδελφό μου, την Υπουργό Δικαιοσύνη, την κυρία Έριξον, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις οι οποίες απευθύνθηκαν προς ε, το άτομό μου. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτή που κάνετε για το Σέγγεν. Και όντω η Προεδρία της Φιλανδίας είναι στη φάση αναζήτηση λύσεων για τους εσωτερικούς ελέγχους. Θα μπορούσαν ενδεχομένω να υπάρχουν ε, πρόσβαση και προσφυγή στους αστυνομικούς ελέγχους, ε, σε λύσεις που μας προσφέρει η τεχνολογία. Σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα, εδώ προφανώς υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο ε, βρίσκεται στη βάση όλων των δράσεών μας. Επίσης, υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο, όπω για παράδειγμα οι επιστροφέ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε τι δράσει μα σε συνεργασία με τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Θα πρέπει λοιπόν όλε αυτέ οι αποφάσει να υλοποιηθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η Φιλανδία θα υποβάλει σχετικέ προτάσει προ την κατεύθυνση αυτή για να δούμε πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ελεύθερη κυκλοφορία και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά την ασφαλειά μα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τώρα. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό. Εδώ είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε πόρους, χρειάζεται να έχουμε ικανότητα αντίδρασης και χρειάζονται λύσεις οι οποίες να μπορούν να κινητοποιηθούν ε, γρήγορα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη διατηρήση της ε, τάξης. Θα πρέπει οι εθνικές αρχές να μπορούν να καταπολεμούν τις ε, τρομοκρατικές ε, δυνάμεις και μάλιστα με ταχύτητα μεγάλη. Να υπάρχουν λοιπόν πόροι και ικανότητε οι οποίε να μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και να υπάρχει και καλή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να επιταχυνθούν ε, οι διαδικασίε ανταλλαγή πληροφοριών και να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση επίση η επικυριαρχία τη κάθε χώρα. Και προφανώ να έχουμε υπόψη μα ότι αυτό επηρεάζει όλε τι πτυχέ τη ζωή μα. Και τίθεται προφανώ το θέμα τη ε, ελευθερία έκφραση. Ε, οι ομιλίε μίσου, οι ευρετικέ απειλέ κατά τη δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια τη ε, Προεδρία μα, επιμένουμε ιδιαίτερω στη διάσταση του κράτου δικαίου. Σε ό,τι αφορά θέματα ελευθερία έκφραση, ελευθερία τύπου, όλα τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ένα σημείο κλειδί ελευθερία έκφρασης. Θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και η λογοδοσία, η υπευθυνότητα. Αυτά πάνε χέρι-χέρι. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο γίνονται συζητήσεις ό,τι αφορά και παράδειγμα προμηθευτές παρόχους ε, ε, διαδικτύου, Facebook, Twitter, ε, πλατφόρμες, όλοι αυτοί έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνη που τους αναλογεί. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συντονιστούν, θα πρέπει να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να γίνει σεβαστή η ελευθερία έκφρασης, λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει και η ευθύνη, η λογοδοσία. Επίσης, για την παράταση του PNR, κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Η γενική ιδέα είναι η εξή. Όπως ξέρετε, οι τρομοκράτες, οι εγκληματίε χρησιμοποιούν διάφορους διάβλου. για την τρομοκρατία λοιπόν και τα... την ε, εγκληματικότητα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συλλογή στοιχείων PNR. Θα πρέπει λοιπόν μαζί τα κράτη-μέλη να βρουν κοινέ ευρωπαϊκέ λύσει και κατά τη διάρκεια τη ευρωπαϊκής ε, της Προεδρία μα θα αναζητήσουμε διάφορου τρόπου που θα μπορούσαν να μα εξασφαλίσουν αυτή την ε, προστασία, παράλληλα με προστασία και τη ε, ιδιωτικής ζωής των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο λοιπόν θα αποφανθεί για τη συλλογή δεδομένων PNR θα δούμε κατά πόσον θα υπάρχει συλλογή δεδομένων και για άλλους επιβάτες πέρα από τους αεροεπιβάτες και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά σε οικονομικό και νομικό επίπεδο. Και τι δυνατότητε υπάρχουν από πλευράς ε, τεχνολογικής. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει ε, που απευθύνθηκαν προ εμένα. Οι υπόλοιπε ερωτήσει έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιο τη Υπουργού Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ λοιπόν να τι απαντήσω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Παρακαλώ, συνάδελφε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 So, Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, της διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεραιότητες διαχείρισης πληροφοριών της Europol για το 2019. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον κύριο Λούις ε, Ντεουσέβιο Ράμος που είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της ε, Ευρωπόλ για τις ε, επιχειρησικές ικανότητες και τον κύριο Άνση Κάγκας που είναι επικεφαλής του προγράμματος UMF3 της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φιλανδίας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ράμος για 10 λεπτά το πολύ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ε, ομάδας ε, Κοινού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Χαρά μου που έχω την ε, ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες για το 2019 να συστηθώ. Είμαι ο, ο Λουίς Εσέβιο Ράμος, ε, αναπληρωτής ε, διευθυντής ε, για ζητήματα επιχειρησιακών ικανοτήτων και διαχείρισης πληροφοριών. Στη στρατηγική της Europol 2020 συν η διαχείριση πληροφοριών έχει προβεβλημένο ρόλο για τον οργανισμό μας. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχει στα χέρια της η Ευρωπόλ. Η διαχείριση λοιπόν αυτών των πληροφοριών βρίσκεται στον πυρήνα των ε, δραστηριοτήτων μας. Και η διαχείριση αυτή δεν είναι μόνο μια υποστηρικτική διαδικασία. Είναι μέρος του DNA του οργανισμού μας, η διαχείριση των πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαχείριση των πληροφοριών για έναν οργανισμό όπως είναι η Ευρωπόλ. Η προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στην Ευρωπόλ όσον αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών είναι μια πρακτική προσέγγιση. Θέλουμε να, να διαθέτουμε τις σωστές πληροφορίες στους σωστούς ανθρώπους στη σωστή στιγμή. Όπως βλέπετε πρόκειται για μια πρακτική προσέγγιση η οποία ε, ωφελεί τους αξιωματούχους τη επιβολής του νόμου ώστε εκείνοι να έχουν τις καλύτερες δυνατέ πληροφορίε τη στιγμή που τις χρειάζονται. Ο ορισμός μας λέει ότι θέλουμε να, να βρίσκονται οι σωστές πληροφορίες στις, στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου για προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Μιλάμε για την καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παντού για όλα αυτά, για αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε πληροφορίες. Και το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε γίνεται, είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και διευρυνόμενο πεδίο. Εδώ στη διαφάνεια βλέπετε τη σημασία που έχει η ε, διαχείριση πληροφοριών από την ε, Europol. Έχουμε πάνω από 10.000 χρήστες που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών μας. Έχουμε 10.000 χρήστες για, του συστήματος της Ευρωπόλ για τη διαχείριση των ε, ε, πληροφοριών μας, όπου μπορεί να κάνει κανείς αναζήτηση, επεξεργασία. Για τους σκοπούς αυτούς έχουμε αναπτύξει και μια διεπαφή που ε, έχει το όνομα Quest, που διευκολύνει τα κράτη-μέλη στην αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9.000 χρήστες στην Ευρώπη του συστήματος αυτού. Τρίτον, έχουμε το Europol Analysis System, ένα εργαλείο στο οποίο μπορεί κανείς, το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν θέλει εις βάθος πληροφορίες ε, που σχετίζονται με εγκλήματα διεθνούς χαρακτήρα. Και τέλος υπάρχει και η πλατφόρμα της Ευρωπόλ για εμπειρογνώμονες. Εκεί έχουν πρόσβαση και άτομα με ε, ευρύτερες αρμοδιότητες. Δεν υπάρχουν εδώ ποινικέ πληροφορίες ε, προσωπικές. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, ανοιχτή και στην έρευνα και στον ιδιωτικό τομέα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16.000 χρήστες αυτής της πλατφόρμας. Οι σημαντικότερες προτεραιότητες διαχείριση ε, πληροφοριών εμφανίζονται εδώ σε αυτή τη διαφάνεια. Πρώτη είναι η διευκόλυνση τη ανταλλαγή πληροφοριών, η κοινή χρήση γνώσεων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αρχών τους. Δεύτερον, η δημιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση της αναζήτησης, της διασταύρωσης και της διαχείρισης δεδομένων. Τρίτη προτεραιότητα, συμβολή του οργανισμού ε, στην ε, ανάγκη ε, εξέβρεσης λύσεων διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γεωγραφικά, αλλά και από άποψη πλήθους ατόμων, οι ανάγκες τις οποίες αντιμετωπίζει ο οργανισμός είναι διαρκώς αυξανόμενος. Με δεδομένο αυτό, βλέπετε εδώ στην ε, δεξιά πλευρά της διαφάνειας την αναλογία ζήτησης και ε, προϋπολογισμού. Η ζήτηση που έχουμε από τα κράτη-μέλη ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός που έχουμε για τεχνολογία πληροφορικής στην Ευρωπόλ είναι 23 εκατομμύρια και ο μεγαλύτερος, ε, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του προϋπολογισμού ε, πηγαίνει σε ε, λύσεις βιωσιμότητας, 19 εκατομμύρια συγκεκριμένου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, η Ευρωπόλη έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στη ζήτηση ε, από τα κράτη-μέλη. Στη διαφάνεια αυτή και στην επόμενη θα σας δείξω τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί και που βρίσκονται ε, προς το προς το τέλος τους. Πρώτον, για το ΣΥΕΝΑ. Έχουμε αναπτύξει νέες διασυνδέσεις με την Γεωργία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων. Δεύτερον, όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ, έχουμε αναπτύξει βελτιώσεις των επιδόσεων χάρη στην αναβάθμιση των τεχνικών στοιχείων αυτής της πλατφόρμας. Και επίσης έχουμε επιτύχει βελτιώσεις όσον αφορά τη διαδικασία αναζήτησης και διασταύρωσης αποτελεσμάτων. Στο Quest το συνδέουμε ε, αυτό το σύστημα με την ε, υψηλής προστασίας υποδομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε έξι χώρες. Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετωνία, Πολωνία και Ρουμανία. Και εκεί επίσης έχουμε εισαγάγει έναν βελτιωμένο αλγόριθμο αναζητήσεων. Όσον αφορά την, ε, το Identity and Access Management, έχουμε ε, δημιουργήσει μια κεντρική ταυτοποίηση επαλήθευση στοιχείων. Κάτι που μας έχει βοηθήσει στο να ε, μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις ε, ικανότητες υποβολής εκθέσεων που έχουμε. Επίσης, έχουμε εγκρίνει στην Ευρωπόλ έναν οδικό χάρτη τον Μάιο του 2019 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Με αυτόν τον οδικό χάρτη θέλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που είναι ενδιαφέρουσες για την Ευρωπόλ με σκοπό να τροφοδοτούν τον οργανωτικό μας σχεδιασμό. Επίσης, αναπτύσσουμε την άμεση πρόσβαση στο σύστημα VIS. και το ΣΥΣ2. Όσον αφορά την ε, αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτή την υποδομή. Για, την αυτόματη, για το σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης βιοματρικών στοιχείων, ρόλος ε, του οργανισμού μας είναι να τροφοδοτεί την Κομισιόν με εμπειρογνωμοσύνη ε, για την ε, επόμενη γενιά Prüm. Όσον αφορά το Universal Messaging Format, το UMF, συμμετέχουμε ε, ενεργά σε δραστηριότητες προγραμματικές στα κράτη-μέλη με σκοπό την συγχώνευση του C1 και του Quest. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας για το 2019. Και θα ήθελα να σας, ε, να σας παρουσιάσω και τις προτεραιότητες του 2020. Πρώτον, έχουμε τις ε, προτεραιότητες ε, των κρατών μελών όσον αφορά τον οδικό χάρτη για την διαλειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ προσφέρουμε το ΣΥΕΝΑ για αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Δεύτερον, απαντούμε, μάλλον επεκτείνουμε το σύστημά μας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε τις αναλυτικές μας ικανότητες και στον τομέα της υπολογιστικής διερεύνησης εγκλημάτων. Και τρίτον, θέλουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα των ε, παραπομπών του διαδικτύου της ε, κοινή ε, χρήσης γνώσεων μέσω της αξιοποίησης των πλατφορμών που έχουμε φτιάξει και ε, την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων και τις σχετικές διαδικασίες που έχουμε αναπτύξει στον οργανισμό μας. Αυτά από πλευράς μου και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Thank you. very pleased to give the floor. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής από τη Φιλανδία έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε η Πρόεδρος, είμαι ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Συνόρων της Φιλανδικής Αστυνομίας. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι το μέλλον της αυτοματοποίησης στα πλαίσια της ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών θέλουμε η συζήτηση αυτή να μπει σε ένα στρατηγικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ένα ευρύτερο επίπεδο που ξεπερνά την εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Και είναι σημαντικό που ήρθε εδώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Θα χρησιμοποιήσω το UMS3 σαν βασικό θέμα εδώ βλέπω ότι έχουμε την φυσική συνέχεια της προσπάθειας την οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε καταφέρει. Στην παρούσα φάση η κατάσταση με την Europol και τα στοιχεία από πλευράς κρατών μελών τα οποία έχει στη διάθεσή της προβλέπεται από τον κανονισμό της Europol, ιδιαίτερα για δεδομένα τα οποία δίδονται για διασταυρώσεις στοιχείων, Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος για τα κράτη-μέλη. Έχουμε επίσης άμεση πρόσβαση και σε άλλου είδους δεδομένα, θεματολογικά και στρατηγικά. Η άμεση πρόσβαση, όπως είπα, προβλέπεται από τον κανονισμό της Europol Ο ισχύων κανονισμός λέει ότι η Europol έχει ε, ένα δεδομένο σύστημα ενημέρωσης, πληροφόρησης, αλλά σε επίπεδο τεχνικό τα συστήματα τα οποία υπάρχουν αντιμετωπίζονται με τμηματικό τρόπο από τα διάφορα κράτη-μέλη εκεί όπου κρατώνται μάλιστα στοιχεία και δεδομένα για διασταυρώσεις. Ήδη έχουμε λοιπόν άμεση ε, πρόσβαση στο EIS της Europol από το ε, βασικό interface, το κοινό interface που χρησιμοποιούν όλες οι ιδιοκτικές υπηρεσίες. Έχει ενδιαφέρον για, ε, για πολίτες όπως τους Φιλανδούς να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα συστήματα αυτά. Εμείς αντιπροσωπεύουμε το 69% όλων των ε, ερευνών EIS το 2018. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και αποδεικνύεται νομίζω ότι έχουμε καλές διαδικασίες και χρήσιμες διαδικασίες. Το UMF3 έχει σαν στόχο την αυτοματοποίηση της εισόδου και της κατάθεσης ερωτημάτων. Η δυνατότητα αυτή, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ονομάζεται Quest και θα πρέπει να είναι σε πιλωτικό στάδιο και βασίζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η πολύ υπεύθυνη γι' αυτό εξ αρχής. Το θέμα είναι να καταστήσουμε ικανούς τους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές ενημέρωσης από τον ίδιο υπολογιστή μέσω μίας κατάθεσης ερωτήματος έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση και στα εθνικά δεδομένα που κατέχει η Europol, αλλά και HISII και γενικότερα και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες μορφές δεδομένων της Europol. Το Quest έχει σαν στόχο να είναι ένα τμήμα του τοπίου διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ε, ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Θύρας Διερεύνησης, του ESP. Να υπογραμμίσω εδώ ότι η Φιλανδική Προεδρία στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουν γίνει σε τεχνικό επίπεδο λέγει ότι βασικός στόχος είναι η απλούστευση του τρόπου χρήσης για τον τελικό χρήστη. Έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να είναι ικανός να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία έχει δικαίωμα να ενημερώνεται. Είναι κάτι το οποίο θα γίνεται ελπίζουμε στο μέλλον, αλλά πολιτικά και νομικά κάτι τέτοιο δεν είναι διασφαλισμένο σήμερα. Όπως είπα, στην πρώτη φάση η λειτουργία του Quest θα στηρίζει ερωτήματα στο κομμάτι EIS του συστήματος και θα δίδει πληροφορίες στα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν ε, ευρέως τα δεδομένα τα οποία έχει αποθηκευμένα η Europol. Έτσι έχει η κατάσταση στην παρούσα φάση. Ε, οι πληροφορίες και τα δεδομένα από το EIS με ε, βάση το interface το αρχικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι κάτι το οποίο λειτουργεί καλά. Το επόμενο στάδιο είναι ότι ο κανονισμός για την Europol ε, πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη μία πρόσβαση hit-no-hit στο αναλυτικό σύστημα, το σύστημα ανάλυσης της Europol ένα διαφορετικό επίπεδο δεδομένων εδώ. Εδώ υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία έχουν σαν στόχο τη λειτουργική ανάλυση. Αυτό θα γίνεται όχι άμεσα αλλά μέσα από τη μέθοδο hit-no-hit. hit no hit Θα υπάρχει δηλαδή εκ των προτέρων έλεγχος για το αν αυτός ο οποίος καταθέτει το ερώτημα έχει δικαίωμα στην χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών. Αυτό το οποίο λοιπόν προβλέπεται και αυτό το οποίο ελπίζεται είναι ότι όταν αυτή η δυνατότητα καταστεί πλήρως λειτουργική τότε θα βελτιωθούν οι δυνατότητες των κρατών μελών για την χρήση των στοιχείων. Θα είναι ένα σύνολο στοιχείων το οποίο δεν θα είναι απλά προσβάσιμο αλλά θα λειτουργεί και αναλυτικά. Οπότε θα έχουμε πληρέστερες αναλύσεις και συνεπώς ανάγκη από λιγότερα στοιχεία. Θα πρέπει να κατανοήσετε εδώ ότι Έχουμε ήδη κάποια μέσα πρόσβασης αυτών των δεδομένων, αλλά η πρόσβαση αυτή είναι αργή, ενώ η λειτουργία αυτή νομίζω ότι θα μας θα διευκολύνει ιδιαίτερα σε επίπεδο ταχύτητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν τις οποίες έχουμε, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν και ανάλογα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους εθνικούς πόρους, θα έχουμε μια δυνατότητα hit no hit τουλάχιστον στα πιλωτικό επίπεδο ήδη από το 2020 και αναφέρομαι μόνο στο hit no hit. Τελειώνοντας την παρουσίασή μου. Νομίζω ότι αυτά όλα θα επιταχύνουν την πρόσβαση των κρατών μελών στα στοιχεία και τα δεδομένα της Europol θα επιτρέψουν τη βελτίωση και τον πολλαπλασιασμό των εθνικών αναλυτικών έρευνών. Το όφελος δηλαδή, ε, το προβλεπόμενο θα είναι όταν πάνε όλα καλά, ε, πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Και τον κύριο και τον κύριο Κάγκα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα και έχουμε λίγο χρόνο πρωτού ε, κάνουμε διάλειμμα ε, για καφέ στι 10.30. Έχουμε κάποιε ερωτήσει λοιπόν. Ε, έχουμε χρόνο για κάποιε ερωτήσει και απαντήσει. Όποιο θέλει να πάρει το λόγο. Αν θέλετε να κάνετε γραπτές ερωτήσεις ή μάλλον να κάνετε ερωτήσεις για τα διάφορα τμήματα της παρουσίασης μας. Δύο λεπτά έχει ο καθένας χρόνο και μετά θα ακούσουμε και τις απαντήσεις. Και από τον κύριο Εουσέβιο και από τον κύριο Κάγκας. Η κυρία Κορνέλη. No? Yes, please. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνούμε δύσκολους ε, καιρούς με μεγάλες προκλήσεις και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Όπως ξέρετε, η Ιταλία έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό συγκεκριμένη υποστήριξη, βοήθεια, γιατί τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι Ιταλικά και τα Ιταλικά σύνορα είναι Ευρωπαϊκά. Χρειάζεται λοιπόν ένα καινούριο σχέδιο ε, δράση, το οποίο θα προβλέπει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μετά των δύο σωμάτων για να υπάρχει καλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς προχωράει αυτό το project. Θα σας υποστηρίξουμε λοιπόν με τις κοινέ αυτές ε, λύσεις και χάρη στην ε, αυτή συνεργασία σε ό,τι αφορά και θέματα κλίματος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και μια δεύτερη... Ο κύριος Μύρα τους από την Κύπρο ζητάει το λόγο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας στο Βουκουρέστι έγινε αναφορά στη δημιουργία ενός εντός του τρέχοντος έτους ενός ε, Travel Intelligence Center της το οποίο θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην επιχειρησιακή και στρατηγική χρήση των πληροφοριών και των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ταξίδια τα οποία προέρχονται από το Αρχείο Ονομάτων Επιβατών. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης αυτού του κέντρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκόφωτ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα ο κύριος Κάγκας να μας διευκρινίσει ένα αριθμητικό στοιχείο που ανέφερε στην παρουσίαση του. Η Φιλανδία ανέφερε είναι η πρώτη σε ό,τι αφορά ε, την αναζήτηση στην ε, Europol. 69 αναφέρεται ως αριθμητικό στοιχείο. Θα ήθελα μια, μια επιβεβαίωση για το αριθμητικό στοιχείο αυτό, αν στέκει όντω. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μάντισον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ήθελε να θέσει ένα θεμείο. Ευχαριστώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε και αντιδράσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούμε διάφορες ιστορίες για τη συνεργασία στη Europol. Φαίνεται ότι υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, σε ό,τι αφορά τη χρήση της λειτουργίας της Europol για την ε, εξασφάλιση της ασφάλειας. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα σε κάποιες χώρες οι οποίες δεν πολύ συμμετέχουν στα της Europol και σε κάποιες περιπτώσεις ε, αντιμετωπίζονται προβλήματα σε ό,τι αφορά την αστυνομική συνεργασία, σε ό,τι αφορά α, θέματα τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Από πλευράς της Φιλανδίας, λοιπόν, τι αίσθηση έχετε, χρειάζεται και να αλλάξετε συνεργασία με τους γειτονές σας, με την Εστονία, τη Σουηδία, όταν ζητάτε στοιχεία, τα λαμβάνετε αυτόματα, γρήγορα, ή αντιμετωπίζετε προβλήματα σε κάποιες χώρες για κάποιους λόγους, σε κάποιες περιφέρειες όπου υπάρχουν προβλήματα. Τι πιστεύετε και τι χρειάζεστε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε η πιο ενεργή χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο. Ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους δύο ομιλητές, τους δύο προσκεκλημένους μας, για να απαντήσουν. Κύριε Σεουσέβιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Με την άδειά σας θα απαντήσω στις πρώτες δύο ερωτήσεις. Ο κύριος με στις δύο επόμενες. Όσον αφορά την συνεργασία Ευρωπόλ Frontex, ε, είναι πράγματι ανάγκη να ενισχυθεί αυτή ε, με νέους κανόνες. Η συμμετοχή συνεργασίας της ε, Ευρωπόλ είναι η αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών. Οπότε, Συμβάλλουμε στους ελέγχους που γίνονται επί τόπου και η συμμετοχή μας γίνεται πάντοτε κατόπιν ε, αιτήματο των τοπικών ερχών. Ανάλογα με τη χώρα, Ιταλία και Ελλάδα είναι οι χώρες από τις οποίες υπάρχουν οι περισσότερες ε, τέτοιες αιτήσει, τα περισσότερα τέτοια αιτήματα ποτέ δεν παρεμβαίνει η Ευρωπόλα αυτεπάγγελτα αν θέλετε, πάντοτε ενισχύει τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου υπό την καθοδήγηση βεβαίως των Ιταλικών και Ελληνικών αρχών. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, για το πρόγραμμα ΕΤΙΑΣ, η συμμετοχή της Ευρωπόλ είναι να συμβάλλει στους ελέγχους όταν το σύστημα πια θα αναπτυχθεί, να διασταυρώνει τις πληροφορίες που προέρχονται από την κεντρική μονάδα του ε, που θα δημιουργηθεί από το Frontex και τον EU Lisa. Η εντολή μας λοιπόν είναι να προσφέρουμε πληροφορίες που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλης στην κεντρική μονάδα του ΕΤΙΑΣ και θα γίνεται διπλός έλεγχος. Επίσης, συμμετέχουμε στην, στον κατάλογο παρακολούθησης που θα καταρτιστεί στον οργανισμό μας ε, σε συνεργασία με, τον, με την Frontex και την EU ε, Lisa. Αυτή τη στιγμή ε, αξιολογούμε τον αντίκτυπο που θα έχουν οι πρωτοβουλίες αυτές όσον αφορά τις εργασίες του οργανισμού μας. Πρέπει να σας πω ότι θα, πρέπει, ότι θα υπάρξουν σημαντικότατες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός μας λόγω του αριθμού των ε, ετοιμάτων που θα λαμβάνουμε και ε, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα πρέπει να είναι μια ε, λειτουργία, μια υπηρεσία που θα παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει ο οργανισμό μας πολύ υψηλές προκλήσεις. Γι' αυτό και ε, κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να παρέχει αυτή την υπηρεσία στις εθνικές αρχές. Αυτά νομίζω ότι απάντησα στα ερωτήματά σας και με την άδειά σας ε, κύριε Κάγκας. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση είναι ναι. Πράγματι, το 2008 το 69% των ε, ετοιμάτων EIS ε, ε, έγιναν από την Φιλανδία. Είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός, πράγματι. Όμως, για να σας ε, περιγράψω τη συνολική εικόνα, μιλάω για τα αιτήματα, όχι για τον συνολικό όγκο των παρεχόμενων πληροφοριών γιατί το μεγαλύτερο όγκο των πληροφοριών τον παρέχουν μεγάλες χώρες και όχι χώρες όπως η Φιλανδία. Ας μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Και ξαναλέω, μιλάμε για τα στατιστικά στοιχεία του 2018, τα περσινά. Φαίνεται ότι το ποσοστό μας φέτος μειώνεται και όχι αυτό δεν συμβαίνει διότι μειώνουμε τα αιτήματά μας, αλλά γιατί αυξάνουν άλλες χώρες τα δικά τους αιτήματα. Η τάση λοιπόν νομίζω ότι είναι θετική. Σχετικά με το ερώτημα για τη συνεργασία πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Πράγματι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπόλ. Κάποια κράτη-μέλη το κάνουν πιο αποτελεσματικά από άλλα. Μετά όμως υπάρχει και το ζήτημα της διμερούς συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Και το ερώτημα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι αν ε, υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κατηγορηματικό όχι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μας είναι ομαλή, πάντοτε στη βάση του ε, των ερωταπαντήσεων και το ποιος έχει δικαίωμα να μάθει τι. Και όταν υπάρχουν προβλήματα τότε συνήθως αυτά οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα, δεν είναι συστημικές ε, οι αιτίε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτήν την διάκριση. Εγώ δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθώ για τη συνεργασία μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Πρόεδρος, έχω λάβει άλλο ένα αίτημα. Από την κυρία Ευελίνα Εινελόμα από την φιλανδική αντιπροσωπεία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες που έχουμε μαζί μας σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση πληροφοριών, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή σκηνή, στο διεθνές στερέωμα, ή σε υπήρους εκτός της Ευρώπης. Και ε, αναρωτιέμαι μήπως έχουμε μείνει πίσω ε, όσον αφορά τη χρήση ε, τεχνολογιών διαχείρισης πληροφοριών ή θα μπορούσατε να πείτε ότι βρισκόμαστε στην πρωτοπορία. Ευχαριστώ. Κύριε Κάγκας, πρώτον, Από εθνική και ευρωπαϊκή σκοπιά θα έλεγα ότι είμαστε ηγέτες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν μπορώ να ξέρω πώς ακριβώς ρυθμίζεται η εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή στις χώρες της Νοτιοαμερικής ή της Αφρικής, της Ασίας. Όλα αυτά προφανώς δεν μπορώ να τα ξέρω. Όμως έχω πολύ έντονα την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τη συνεργασία μας με τον έξω κόσμο, από τη δική μου σκοπιά πάντοτε, που είναι η ανταλλαγή διεθνών πληροφοριών ε, σε ποινικά ζητήματα, ε, πρέπει να σας πω ότι εμείς βασιζόμαστε πάντοτε στην Ιντερπολ. Ο κύριος Ευσέβιο. Ευχαριστώ. Να απαντήσω κι εγώ στα ερωτήματα αυτά. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις που διαπιστώνουμε είναι η χρήση ε, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης μηχανικής. Εμείς ε, παρακολουθούμε στενά το ζήτημα αυτό με τη βοήθεια των αναλυτών της Ευρωπόλ. Αυτό σχετίζεται και με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας προκειμένου να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα μηνύματα από τα κράτη-μέλη και προκειμένου να διευκολύνουμε και να ε, ε, επιταχύνουμε το χρόνο εντός του οποίου το προσωπικό της Ευρωπόλ δίνει απαντήσεις στα διάφορα αιτήματα δηλαδή που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει το προσωπικό μας, για παράδειγμα. Αυτό ε, συμβαίνει, για παράδειγμα, με τα συστήματα. Υπάρχουν συστήματα τα οποία λαμβάνουν μηνύματα, επεξεργάζονται τουλάχιστον σε ένα, σε ένα πρώτο στάδιο το περιεχόμενο, τον τίτλο, την κατηγορία του, του μηνύματος και μετά κατηγοριοποιούν τα μηνύματα αυτά και τα διαβιβάζουν μεταβιβάζουν σε, στους ε, αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι να τα επεξεργαστούν. Όσον αφορά τα υπερσύγχρονα εργαλεία προκειμένου να λαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που λαμβάνουμε. Για παράδειγμα, ε, στην, στην, ε, στα εγκληματολογικά ζητήματα, για παράδειγμα, στα ζητήματα διερεύνησης εγκλημάτων, ο όγκος που λαμβάνουμε είναι τεράστιος όγκος των πληροφοριών και των δεδομένων. Βίντεο, για παράδειγμα, ε, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και παιδικής κακοποίησης. Οπότε χρειάζομαστε πάρα πολλούς πόρους και πάρα πολύ χρόνο για να επεξεργαζόμαστε. Για το ε, ε, υπολογιστικό νέφος εμείς δεν το χρησιμοποιούμε λόγω περιορισμών που προβλέπονται από την νομοθεσία. Έχουμε συστήματα στην ε, Ευρωπόλ που καθιστούν συγκεκριμένε πληροφορίε και πολλέ κατηγορίε ε, πληροφοριών ω εμπιστευτικέ και γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε υπηρεσίε υπολογιστικού νεφου. Ευχαριστώ κύριε Ουσέβιο, Διευθυντή τη Ευρωπόλ, εκτελεστική, εκτελεστική Διευθυντή και τον κύριο ε, από την ε, αστυνομία τη Φιλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τις απαντήσεις σας. Είναι προφανές ότι η διαχείριση πληροφοριών είναι ένα ζήτημα ολοένα και πιο σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τον του, του αυξανόμενου όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών. Οπότε είναι απαραίτητο να, να ε, συμμορφωθεί η διαχείριση των πληροφοριών με τις αρχές των θεμελιωδιωδών δικαιωμάτων και τις προστασίες των προσωπικών δεδομένων. Πάμε σε διάλειμμα για καφέ. Όμως, να σας πω από τώρα ότι μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τον εσωτερικό κανονισμό και τις σχετικές τροποποιήσεις επί αυτού. Υπάρχουν διάφορες συμβαστικές προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί εκείνοι που έπρεπε να το κάνουν. Χρειάστηκε πολλή δουλειά και πολλής χρόνος για να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα πρότεινα λοιπόν ότι εκείνοι που θέλουν να ε, προσθέσουν κάτι σε σχέση με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στον εσωτερικό κανονισμό, σας παρακαλώ να τις καταγράψετε αυτές τις προσθήκες ή αλλαγές σας και να τις ε, συμπληρώσετε εδώ στα έντυπα που έχουμε στη διάθεσή σας, ώστε να ξέρουμε μετά το διάλειμμα ποιος ε, θέλει να προσθέσει τι στις συμβαστικές προτάσεις που έχουν επιτευχθεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έγιναν. Πάμε για καφέ και τα ξαναλέμε.

colleagues. Dear colleagues, now we are just continue. Please. Συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. We continue our debate on the revision of... Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ε, ε μεταρρύθμιση των κανόνων και των διαδικασίων και Χτες είχαμε συζήτηση για τη συμμετοχή της Δανίας, ακούσαμε την παρουσίαση των αντιπροσωπείων. Σε ό,τι αφορά την κανονισμό του TBST, αποφασίστηκε με ομοφωνία. Να σας υπενθυμίσω και τη σχετική γνωμοδότηση που διευκρινίστηκε και χθε ότι η χθεσινή συζήτηση και η σημερινή συζήτηση θα σημάνει και το τέλος της διαδικασίας για την μεταρρύθμιση του κανονισμού. Οι συμπρόεδροι θα δώσουν αναφορά στη διάσκεψη των πρόεδρων της, των κοινοβουλίων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας μετά τη συνάντησή τους τον Απρίλιο. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση λοιπόν τώρα. Να δώσουμε το λόγο στα μέλη που ζήτησαν να μιλήσουν για δύο λεπτά κατά το όριο το κείμενο από την ε, Φιλανδική Αντιπροσωπεία. Κυρία Πόρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρώτα. Εξ ονόματος της Φιλανδικής Αντιπροσωπείας θα ήθελα να παρουσιάζω μία τροπολογία για το άρθρο 5. Την έχετε λάβει και γραπτά στο, στα έντρανα σας, να τη διαβάσω για το άρθρο 5, αρωπή. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ε, κανονισμού για το Europol, οι συμπρόεδροι θα παρουσιάσουν το GPS, θα εκπροσωπούν το GPSE στο Διοικητικό Συμβούλιο του Europol ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο πρόεδρος της Τρόικα θα συμμετέχει στις διαδικασίες για την προετοιμασία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι θα αναφέρουν στο GPSC τι έγινε μετά από κάθε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα παρουσιάσουν τα βασικά πορίσματα εγγράφως. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέλκον από την Ολλανδία. Πρόεδρε, χτες η αντιπροσωπεία GPSS Κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πολύ χρήσιμη για τις ε, τροπολογίε για τον κανονισμό. Διάφορες αντιπροσωπείε και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάστηκαν πολύ σκληρά για να προετοιμάσουν ε, τις τροπολογίε αυτές και να τι καταθέσουν. Και από το έγγραφο σύνοψη τη ε, Προεδρία, όπου γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των τροπολογίων και από τη χθεσινή ανταλλαγή απόψεων, η Ολλανδική Αντιπροσωπεία εξαγάγει ο συμπερασμά ότι δεν θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ενδεχόμενη αλλαγή του κανονισμού. Και επιπλέον δεν είχαν όλε οι αντιπροσωπείε την ευκαιρία να εκφραστούν επί του περιεχομένου ή επί τη διαδικασία, γιατί δεν υπήρχε χρόνος ε, στην διάρκεια των ε, διασκέψεων. Γι' αυτό λοιπόν η Ολλανδική Αντιπροσωπεία θα πρότεινε ένα ερωτηματολόγιο. Να ρωτήσουμε όλες τις αντιπροσωπείες να απαντήσουν γραπτά σε ό,τι αφορά τις ε, υποβλήθεις ε, σε τροπολογίες ε, και τις πρόταση της Φιλανδικής Αντιπροσωπείας και επίσης οι αντιπροσωπείες να μας πούν κατά πόσον θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με τα τμήματα των τροπολογιών. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο για να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό ο οποίος θα είναι ευρύθμος. Και επίση θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο και να δούμε πώ μπορούν να διατυπωθούν σωστά οι τροπολογίε, οι οποίε ελπίζουμε να εγκριθούν στην επόμενη διάσκεψη. Η Ολλανδική Αντιπροσωπεία καταθέτει την πρόταση αυτή, γιατί πιστεύετε ότι θα είναι πάρα πολύ κρίμα να χωρίσουμε δρόμους χωρίς να έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα προς τα εμπρό. και θεωρούμε ότι αυτό το ενδιάμεσο βήμα με τη μορφή του ερωτηματολογίου θα ήταν κάτι απαραίτητο για να πετύχουμε κάποια πρόοδο και θεωρούμε ότι θα ήταν ωφέλιμο και χρήσιμο για τη συζήτησή μας και θα μπορούσε να συμβάλλει για πιο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας της ομάδας μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And then Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιστόρης από τη Γερμανία. Συνάδελφοι, από γερμανικής πλευράς θέλω επιτακτικά να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια προθεσμία για την υποβολή απαντήσεων. Αν δεν ρυθμίζεται πότε θα πρέπει να δίνονται οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν δοθεί στους συμμετέχοντες ε, είναι ένας μηχανισμός ε, μη, ανα, ε, μη αποτελεσματικός, αναποτελεσματικός. Γι' αυτό και πρέπει εδώ στο Κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε και να το επισημάνουμε με ότι ελήφθη μια σχετική απόφαση ε, με ομοφωνία. Δεν είναι δευτερεύουσα σημασία κάτι τέτοιο. Πρέπει να οριστούν προθεσμίε. Και δεύτερον, ω Υπουργό εσωτερικών Κρατηδίου τη Γερμανία, θα ήθελα να δούμε κάποια στιγμή και τον ιστορικό οργανισμό του Ιουλίσα, για παράδειγμα. Ζήτημα, ζήτημα δικαστήρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακροδεξιά τρομοκρατία. Νομίζω ότι τα θέματα που μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια εδώ μέσα ε, είναι ζητήματα που είναι δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί έξω. Ο, κύριο, ο κύριος Άπολα από την Πολωνία. Uh, Mr. Peters from please. Ο κύριος Πέτρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρώτον, υποστηρίζω την ιδέα ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό σήμερα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο εσωτερικό κανονισμό βεβαίω, το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζω και εγώ, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να τελειώσουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα. Δεύτερον, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπάθησε βεβαίως να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις όπου αυτό ήταν εφικτό. Έλαβα και την πρόταση συμβασμού της φιλανδικής αντιπροσωπείας σχετικά με το άρθρο 5 και θεωρώ ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποδεχθεί αυτό τον συμβασμό με την ελπίδα βεβαίως ότι μπορούμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για άλλα πολύ σημαντικά θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Λέοπαρ από την ε, Σουηδία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις βασικές προτάσεις από τις αντιπροσωπείς της Γερμανίας, Φιλανδίας και της Ρουμανίας για το άρθρο 5. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να υποβάλουμε μια πρόταση σουηδικής αντιπροσωπείας για να αλλάξουμε το άρθρο 6.2 και να εισαγάγουμε μια νέα ειδική διαδικασία η οποία θα επιτρέπει στι αντιπροσωπείε να υποβάλουν προτάσει για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Δημητρίου από την Κύπρο. Ναι, καλή σας μέρα. Είναι όντως πολύ σημαντικές οι τροπολογίες, αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό να τελειώσουμε σήμερα με αυτό το ζήτημα που εκκρεμεί και είμαστε στην πέμπτη σύνοδο και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στο άρθρο 5. Ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και οι τροπολογίες 4 και 5, η μια από την Ολλανδία και η άλλη από την Γερμανία, την Κροατία και την Ρουμανία, εμεί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί ο χρόνο και συμφωνούμε σε αυτέ. Τώρα, σε σχέση με τη συμβιβαστική πρόταση που έχει κατατεθεί σήμερα από τη Γερμανία, την Φιλανδία και την Ρουμανία για το άρθρο 5. Είναι πολύ καλό πιστεύω να επεξηγηθεί σε όλους και ο ορισμός του alternately όπως καταγράφεται στην τροπολογία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε την βασική αρχή πως τα κράτη είναι αυτά που έχουν την εξουσία και είναι αυτά που πρέπει να συμφωνούν ή να διορίζουν αυτό τον εκπρόσωπο. Αν επιλέξουν να είναι εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώς. Επίσης, στην λογική αυτή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε, αφού θα έρχεται πρόσκληση από το Management Board, να προσκαλείται πάντοτε ο εκπρόσωπος της χώρας και να είναι ο, ο Ευρωβουλευτής αυτός που θα είναι ο επιλαχών ή ο, αντικαταστάτης. Ευχαριστώ. Thank you. And then Mrs. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φλωρά από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς υποστηρίζουμε ε, την πρόταση της Σουηδικής Αντιπροσωπείας, το αναφερμένο κείμενο. Θεωρούμε ότι είναι καλή και η ιδέα της ε, Ολλανδικής Αντιπροσωπείας. Να υπενθυμίσω ότι είναι η τελευταία φορά που μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Άπαξ και αλλάξει, μετά θα ισχύει. οι ερωτήσεις είναι το, μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να ασκούμε τον έλεγχό μα. Γι' αυτό και χρειάζεται να ε, εξασφαλιστεί αυτή η περίοδο των έξι εβδομάδων που κατοχυρώνεται στον κανονισμό. Και θα πρέπει να κατευθυνθούν και, όλα τα ερωτήματα σχετικά με το IPAX. Επίσης, ε, να υπενθυμίσουμε ότι ε, ο εσωτερικός κανονισμός ε, είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς με, βάση το οποίο προσανατολιζόμαστε. Χρειαζόμαστε έναν κανονισμό. Ο κ. Μετώνιο από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Η, η γερμανική φιλανδική ε, πρωτοβουλία μας βρίσκει σύμφωνος με μία μικρή τροπολόγηση όμως, η πρώτη φράση μόνο να πούμε ότι σε σχέση με το άρθρο 14 του κανονισμού ο συμπρόεδρος ή συμπρόεδροι μάλλον δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Και θα πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε καλύτερα για ποια περίοδο η αντιπροσώπευση αυτή θα ισχύει. Ευχαριστώ. Από τη Γαλλία. Συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι εδώ και αρκετές συναντήσεις προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε επίπεδο εσωτερικού κανονισμού και θα πρέπει να καταλήξουμε με επιτυχία. Δύο παρατηρήσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λείπει στα πλαίσια της δουλειάς που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι μια βασική προτεραιότητα, δηλαδή τα μέσα για τη διασφάλιση του ελέγχου. Περάσαμε πολύ χρόνο στον εσωτερικό κανονισμό και τους κανόνες του. Σωστό είναι αυτό. Αν χάσουμε όμως το πώς θα κάνουμε τον έλεγχο, γιατί εδώ και πολλούς μήνες το συζητάμε αλλά δεν καταλήγουμε πουθενά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ε, λύση που να ικανοποιεί όλους. Η φιλανδική πρόταση πιθανής μεταβατικής περίοδου μπορούμε να τη στηρίξουμε αλλά υπάρχουν ε, ελλείψεις. Αυτό το οποίο ελείπει σήμερα και συνδέομαι εδώ με αυτά τα οποία είπε και η σουηδική πλευρά είναι η έκτακτη διαδικασία αναθεώρησης, γιατί στον δικό μας κανονισμό δεν υπάρχει αναθεώρηση και συμφωνώ με την Ρουμανία σε αυτά τα οποία είπε. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν σε κάποια στιγμή να προβλέψουμε μία συγκεκριμένη στιγμή όπου με έκτακτο ή τακτικό τρόπο θα προβλέπεται μία απαραίτητη εφόσον υπάρχει η ανάγκη αναθεώρηση. Κατανοώ την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει βήματα προόδου ε, για την Europol. Να μην ξεχνάμε όμως, και αυτό έχει υποθεί επανειλημμένα, ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν έχουν ακόμα προβλεφθεί και οι χρηματοδοτήσεις περνούν και από τα εθνικά κοινοβούλια. Είμαστε μεν πεπισμένοι όλοι για τη δουλειά που κάνει η Ευρωπόλ και για τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό τον οποίο πρέπει να υφίσταται. Δεν μπορούμε όμως να στηρίξουμε το αίτημα αυτό για επιπλέον μέσα αν ο διάλογος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν ε, ε, ολοκληρωθεί χρονικά στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού. Η πρόταση λοιπόν η οποία γίνεται είναι μια πρακτική πρόταση, ενδιάμεση όμως, και το θέμα της αναθεώρησης και πιθανώς των μέσων τα οποία θα χρειαστούν για να υπάρξει έλεγχος επιβάλλεται να βρεθούν από τώρα. ο Ιρλανδός εκπρόσωπος. Διαβάζοντας την αρχική πρόταση από Φιλανδία, Γερμανία και Ρωμανία, βλέπουμε ότι έχουμε τα μέσα ε, στη διάθεσή μας για να δεχτούμε τις προτάσεις αυτές. Υπάρχει ανάγκη για κάποιες ε, διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 14 σαν παράδειγμα στα πλαίσια όμως ε, της παρουσίας δύο μελών για δωδεκάμινη περίοδο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το κράτος μέλος που έχει την Προεδρία δεν θα έχει τον επιπλέον εκπρόσωπο και δεν θα έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει σωστά τα πράγματα. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των αντιπροέδρων οι οποίοι θα εκπροσωπούν διαδοχικά ή και οι δύο μαζί. Και επίσης το θέμα της ψήφου των αντιπροέδρων είναι σημαντικό και θέλουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Έχει σημασία να καταλήξουμε σε μια τελική θέση και σήμερα αν είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να κάνουμε συζητήσεις για θέματα ουσίας σε σχέση με τον έλεγχο τον δημοκρατικό της Europol. Ευχαριστώ συνάδελφε. Να πω στην Ολλανδική Αντιπροσωπεία ότι όλοι είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους οι συμπρόεδροι μπορούν να τα, να υπόψη τους όλα αυτά και να δουν ακριβώς ότι ε, προτάσεις θα κάνουν. Ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να σημειώσουμε μετά από τη μεταφορά όλων αυτών των προτάσεων στους, στην διάσκεψη των Προέδρων. Θα περιμένουμε λίγο. Η Πορτογαλική αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ, λέει η Πορτογαλίδα εκπρόσωπος, για τη συμβιβαστική πρόταση η οποία μας έχει κατατεθεί υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε. Η εναλλαγή είναι μια ιδέα που έχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση γύρω από το θέμα της εναλλαγής. Όταν υπάρχει συνάντηση των αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες, ε, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς συνδυάζεται με την προεδρία την οποία πρέπει να ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια. So, um, another. Uh, Miss Mittag. Κυρία Μιτάκ, από τη γερμανική αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ äh, für das Wort. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Η συζήτηση νομίζω καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποια βεβαιότητα για το πώς θα α, ακολουθηθεί η μελλοντική διαδικασία, τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Δεν μπορούμε να πετύχουμε μια ομοφωνία η οποία δεν υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι σύμφωνα με τις ε, κατευθυντηρίες γραμμές θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη ειδική πρόταση για την ρήτρα αναθεώρησης γιατί δεν θα πετύχουμε συμφωνία εδώ. Παρόλα αυτά όμως το θέμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Ναι, μεν πρέπει να το κλείσουμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και ένα παράθυρο ανοιχτό για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να τα ρυθμίσουμε αυτά. Και οι χώρες ε, τι συμφέροντα έχουν, γιατί όλα αλλάζουν αν ε, κάποια τροπολογία, ναι μεν μπορεί να μην ε, συγκεντρώνει την πλειοψηφία όλων μας, αλλά παρόλα αυτά να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε την πρόταση τη Ιουδική Αντιπροσωπεία να υπάρξει ρήτρα αναθεώρηση, να το σκεφτούμε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση για να δούμε πώ θα πατήχουμε τελικά συμφωνία. Και να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια τη Επιτροπή Γεωργοπόλου. Ευχαριστώ. Tässä useampi kysyi tästä puheenjohtajuudesta vastaan siihen suomeksi. Ευχαριστώ πολύ που θέσατε το ερώτημα αυτό. Θα απαντήσω στα φιλανδικά. Η συμπροεδρία λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Βρυξέλλες των κρατών μελών οι πρόεδροι λοιπόν συμφώνησαν για να αποφασίσουν ποιος θα έχει το ρόλο των αντιπροσώπου. Eli hyvät kollegat. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε διάφορε παρέμβάσει, ακούσαμε τι απόψει των ε, συναδέλφων και όπω διαπιστώσαμε όλοι μα. παραμένουν ακόμα εκκρεμή ζητήματα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικέ απόψει. αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ομοφωνία στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι επ' αυτού συμφωνούμε όλοι. Επί της αξιολόγησης δηλαδή της κατάστασης όλοι είμαστε σύμφωνοι. Eli liittyen nyt sitten Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5. Μιας και δεν υπάρχει ομοφωνία, απορρίπτεται η πρόταση. Ναι. So we continue based on the in the in the να συνεχίσουμε να σας πω ότι τα αποτελέσματα της συζήτησης για τις προτινόμενες τροπολογίες και για τους συμβιβασμούς έχει ως εξή. Να κοιτάξουμε τις τροπολογίες μία προς μία. Τροπολογία 1 από την Ολλανδική ε, Αντιπροσωπεία. 3-3, άρθρο 3-3. Η Τρόικα είναι αντίθετη με την τροπολογία αυτή. Δεν υπάρχει ομοφωνία. για την αλλαγή του κανονισμού και την προσαρμογή αυτού. Τροπολογία 2. Από τη γερμανική αντιπροσωπεία για την ατζέντα των συναντήσεων, άρθρο 4.1. Α. Συμφωνούμε επί τη αρχή με το μεγαλύτερο κομμάτι τη τροπολογία. Παρ' όλα αυτά, διάφορε αντιπροσωπείε εξέφρασαν αντιρρήσει σε, ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλο. Επ' αυτού θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει μια συνένεση. Σε ό,τι αφορά την προτινόμενη αλλαγή όμως του κανονισμού δεν εγκρίθηκε. 3 και 8, τρίτη και 8η τροπολογία από την τσεχική αντιπροσωπεία και από τη Σλοβενία για τη λήψη αποφάσεων στο JBST. αρθρο 1 4.1α και η διάφορες αντιπροσωπείες ήταν ε, κάθετα αντίθετες σε ό,τι αφορά την αρχή της συνένεσης όπως συμφωνήθηκε από την διάσκεψη της πρώτης το 2017. Δεν εγκρίθηκε λοιπόν η προτινόμενη αλλαγή του κανονισμού. Τροπολογία 4 από Bundestag και Bundesrat και από τη Ρουμανική και Κροατική αντιπροσωπεία. Τροπολογία 5. Για το δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων. 5-2. Σύμφωνα. Παράθεση από πριν που έγιναν να βρούμε συμβιβασμό και τις συζητήσεις ε, για τον οδηγό για τα μέλη, σε ό,τι αφορά τι και προφορικές ερωτήσει, ε, δεν πετύχαμε συμφωνία. και έτσι δεν εγκρίθηκε η προτινόμενη αλλαγή του κανονισμού. Τροπολογία 6, 7, 9, 10, 11 και 12 από διάφορες αντιπροσωπείες σχετικά με τον εκπρόσωπο της JPSG στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ, άρθρο 5. Δεν υπάρχει συνένεση. η προτινόμενη αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού δεν εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 του, του Σουηδικού Κοινοβουλίου, τελικές διατάξεις, άρθρο 6. Ούτε εδώ επετέφθη συνένεση επί του άρθρου αυτού, οπότε δεν εγκρίθηκε ούτε αυτή η προτινόμενη αλλαγή του ιστορικού κανονισμού. Αυτά σε σχέση με τις τροπολογίες. Μάλιστα. Ε, υπάρχει μια κούραση από τους συμμετέχοντες μετά από τις μακρές συζητήσεις που έγιναν για αυτούς τους διαδικαστικούς κανόνες, για τον ιστορικό κανονισμό, οπότε καλό είναι ε, και εύλογο να φτάσουμε σε ένα τέλος. Αφού δεν υπάρχει συνένεση, εξακολουθούν να ισχύουν ή κανόνες ως ίσχυαν σχετικά με τη συμμετοχή της Δανίας και την σχετική αλλαγή. Εγκρίθηκε αυτή χτες. Και τίθεται η αλλαγή ε, αυτή σε ισχύ αμέσως. Ξαναμιλά, ξαναλέω ότι αναφέρομαι στην, στους κανόνες που σχετίζονται με την Δανική συμμετοχή. Δυστυχώς δεν φάνηκε να υπάρχει συνένεση στα άλλα ζητήματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία αναθεώρησης του ιστορικού κανονισμού. Γιατί γνωρίζετε ότι καθήκον των συμπροέδρων είναι η λογοδοσία στους ε, Προέδρους των Εθνικών Κοινοβολίων σχετικά με την ε, αλλαγή στον εσωτερικό κανονισμό. Στη βάση αυτών, αυτού του απολογισμού που θα γίνει, οι συμπρόεδροι μπορούν να εξετάσουν περαιτέρω βήματα που θα μπορούσαν να αναλυθούν προκειμένου να επιδεχθεί ε, συνένεση σε πιθανές συμβιβαστικέ προτάσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση που πρέπει να κάνω. Πρωτού περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά τον διορισμό, τον εκπρόσωπο του JSPG στη συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ε, της Ευρωπόλ που συνεδριάζει ε, στη Χάγη, στην έδρα του οργανισμού. Και εδώ επιχειρήθηκε να βρεθεί συνένεση και συμφωνία, έγιναν συζητήσεις, λάβαμε υπόψη μας όλες τις συνεισφορές στη συζήτηση αυτή όμως, όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτών των ε, συζητήσεων, μπορώ να ανακοινώσω ότι δεν υπάρχει έδαφος συνένεσης όσον αφορά την τροποποίηση των ισχυών των ε, κανόνων του ιστορικού κανονισμού. Οι συμπρόεδροι θα συνεχίσουν λοιπόν να εκπροσωπούν το GSPG στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ στις συνεδριάσεις του. Και με αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση που έγινε για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού. Του τουλεχθέντος θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στο τελικό κομμάτι, στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνεδρίασης, συνάντησης. Οπότε, περνάμε στις τελικές παρατηρήσεις. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Ταλβίτιε για να κάνει τις ε, τελικές παρατηρήσεις το κλείσιμο δηλαδή αυτή της συνεδρίασης της Ομάδας Κοινού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Ευχαριστώ αγαπητέ συμπρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή. Ελπίζω ότι οι παρουσιάσεις που έγιναν χθες και σήμερα, οι συζητήσεις που έγιναν χθες και σήμερα, θα φέρουν ένα βήμα πιο κοντά την ομάδα μας στον στόχο τους, δηλαδή την, τον πολιτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Shall I go now? Yeah. So, thank you all. Thank Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας, για την συνεισφορά σας στη συζήτηση, στην ανταλλαγή απόψεων, για όλη τη δουλειά που έγινε, για όλα όσα έγιναν, όχι μόνο στους τελευταίους ε, μήνες, αλλά ιδίω όσον αφορά τον εσωτερικό οργανισμό εδώ και χρόνια. Πολλοί είπατε ότι πραγματικά ήταν ώρα πια να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση και προχωράμε με την ε, θεσμοθέτηση πλέον αυτής της μορφής του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ε, Ευρωπόλ. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αναμφίβολα, που αποδεικνύει και την αξία που έχει η ομάδα μας και δεσμευόμαστε ότι στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση θα ασκούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει τον Μάρτιο του 2020 υπό την αιγίδα της Κροατικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επομένως θα γίνει στην Κροατία. Δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πού, όμως θα διοργανωθεί από κοινού, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Κροατίας. Φυσικά στο μεσοδιάστημα θα βρισκόμαστε σε επαφή με την Ευρωπόλ και θα ασκούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των, των ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και ιδίως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ για τη συμβολή σας στις συζητήσεις που έγιναν. στις ομάδες εργασίας που αποτελούνταν από εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών θα διανεμηθούν σε, όλα, σε όλους τους συμμετέχοντες από το Εθνικά Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας, για τη συνεισφορά σας, για τη δουλειά που κάναμε. Καλό ταξίδι επιστροφής στους εθνικούς βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε την επόμενη φορά στην Κροατία. Γεια σας.